στην Ουκρανία. Ελπίζω <clears throat> ότι ακόμα δεν έχουμε λόγους για σοβαρές ανησυχίες. <clears throat> Ευχαριστώ τον κύριο Μπέλντερ. Ακολουθούει ο κύριος Μέλτσερ για τους μη εγγεγραμμένους. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ξέρουμε όλοι ότι η Ουκρανία είναι μία από τις πιο κοντινές γειτονικές χώρες